Good afternoon. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Και καλησπέρα σας κιόλα. Hi. It's like this. Good afternoon to everybody. Καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε όλοι σε αυτή την συνεδρίαση της νέας θητείας της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κλπ. Και πρόκειται να προεδρεύσω της συνεδρίας αυτής που έχει ως σκοπό να εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής μας. Ε, προεδρεύω εγώ γιατί είμαι η βουλευτήνα που έχει τις περισσότερες αρμοδιότητες στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και στην θητεία επίσης θα είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής. Επομένως, κηρύσω την έναρξη της ε, συνεδρίασής μας και επίσης πρέπει να σας πω ότι πρέπει να εκλέξουμε τα μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής Απασχόλησης και Γενικών Υποθέσεων θα πρέπει να εκλέξουμε πρόεδρο και αντιπροέδρου σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Πρώτα πρώτα, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης. Αυτόν πρέπει να εκλέξουμε. Σας βεβαιώνω ότι υπάρχει απαραίτητη απαρτία. Παρακαλώ τώρα οι πολιτικές ομάδες να προτείνουν τους υποψηφίους τους. Δώ palavra a Patrick Liarric do Guengel. Πατρίκ Λιαρίκ, από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική μας ομάδα θα προτείνει ως υποψήφιο τον Τόμα Έντελ για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο Τόμας Έντελ είχε αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα κατά την τελευταία θητεία ή στην Επιτροπή αυτή. Ήταν δε συντονιστή της πολιτική μα ομάδα σε αυτήν την πολιτική ομάδα αλλά και στη χώρα του τη Γερμανία έχει σημαντική συνδικαλιστική εμπειρία στα εργατικά και εργασιακά και συνέταξε μία σειρά από γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις κατά την προηγούμενη θητεία. Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε. Κύριε ε, θέλει ο υποψήφιος να λάβει το λόγο. Δέχεστε, ναι. Ωραία. Για πέστε μας. Έχετε συμπληρώσει την ε, δήλωση των οικονομικών συμφερόντων. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε άλλη υποψηφιότητα. Επομένω, σα προτείνω να εκλέξουμε διαβοή τον κύριο Χέντελ ως πρόεδρο μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχικώς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, εμπιστοσύνη σας να μου αναθέσετε τα καθήκοντα του Προέδρου. Θα σας μιλήσω στη συνέχεια και για τα, τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από τώρα ότι θέλω να συνεργαστώ ανοιχτά, έντονα και με διαφάνεια με όλα τα μέλη της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή θεωρώ, αυτή την περίοδο, η Επιτροπή μας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και την αλληλεγγύη και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μας για να καταλήγουμε πάντοτε σε καλές λύσεις για τους πολίτες της Ευρώπης. Τώρα, να προχωρήσουμε στην συγκρότηση του Προεδρείου. Θα γίνει τώρα η ψηφοφορία για τους αντιπροέδρους της Επιτροπής αυτής. Συνολικά τον αριθμό είναι τέσσερις. Να ζητήσω λοιπόν τώρα να υποβληθούν υποψηφιότητε για, για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ. Η κυρία Ροντρίγε θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα. Καλησπέρα. Μιλώ εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ως αντιπρόεδρος της ομάδας αυτής και η ομάδα μας θα ήθελε να προτείνει τον εξής συνάδελφο για πρώτο αντιπρόεδρο. Μιλούμε για την Μαρίτα Ούλσκοκ. Την κυρία Μαρίτα Ούλσκοκ. Μαρίτα Ούλσκοκ. Ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Συμφωνεί η κυρία Ολσκούκ με την υποψηφιότητά της. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ε, yes. Um, I... Ναι, αποδέχομαι. Την υποψηφιότητά μου το όνομά μου είναι Ulf Σκούγ. Ωραία. Θα εξασκηθώ πιστεύω μέχρι το τέλος της θητείας θα τα καταφέρω να το προφέρω σωστά. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπομένως υπάρχει συμφωνία. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων έχει υποβληθεί και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια σας όσοι συμφωνείτε. Ωραία. Σας συγχαίρω. Μαρίτα, παρακαλώ μπορείς να έρθεις να καθίσεις δίπλα μου. Ωραία. Άρα προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία για τον δεύτερο αντιπρόεδρο ή την δεύτερη αντιπρόεδρο. Ο λόγος στον Έντουαρτ Κουκάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ προτείνουμε την κυρία Γιαζλοβιέτσκα για τη θέση του δεύτερου του Προέδρου της Επιτροπής. Η κυρία Γιασλοβέτσκα στην προηγούμενη θητεία ασχολήθηκε με πολλά σημαντικά ζητήματα με αποτελεσματικότητα και νομίζω ότι αυτό της ε, προσδίδει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για τη θέση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ντανούτα Γιασλοβιέτσκα. Συμφωνεί η ίδια. Πού είναι. Α, δεν είναι παρούσα. Μου λέει η ομάδα της όμως ότι συμφωνεί με την υποψηφιότητά της, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην, στην ψηφοφορία. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Όχι. Επομένως εκλέγεται η Ντανούτα Γιαζλοβιέτσκα διαβοής. Παρακαλώ τώρα. Ωραία. Και φτάσαμε με αυτό στην ψηφοφορία για τον τρίτο αντιπρόεδρο ή την τρίτη αντιπρόεδρο. Και εδώ έχω πρόβλημα με το όνομα, αλλά θα το ακούσω ε, σε λίγο πώς προφέρεται. Για να Τόμ θα μας πει. Ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων θα ήθελα να υποβάλω υποψηφιότητα για την κυρία Ούλα Τέρνας. Δυστυχώς δεν είναι παρούσα, αλλά έχω μαζί μου μια δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία συμφωνεί και αποδέχεται τη θέση, εάν και εφόσον εκλεγεί σήμερα. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε επίσης και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, όπως προβλέπετε. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Όχι. Άρα προχωρούμε στην ψηφοφορία. Όποιο συμφωνεί με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Δεν υπάρχουν ψήφοι κατά. Επομένω, η κυρία Ούλα Τέρνες εκλέγεται τρίτη αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Δεν είναι παρούσα. Ευχαριστώ πολύ και περνούμε στην ψηφοφορία για την τέταρτη αντιπρόεδρο ή τον τέταρτο αντιπρόεδρο. Η Μαρία Τζοάο Ροντρίγκες ροντριγκε εχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι ως αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχουμε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την υποψηφιότητά μας για τον τέταρτο αντιπρόεδρο αυτής της ε, Επιτροπής. Κάθεται μπροστά μου. Είναι η κυρία Άγνιες Γιονγκέριους. Να τονίσω ότι η υποψήφια μας ότι η υποψήφια μας για την θέση του πρώτου αντιπροέδρου που μόλις εξελέγει είναι ένα εξαιρετικά πεπειραμένο μέλος του κοινοβουλίου μας και τώρα είμαστε στην ευχαριστή θέση να σας ε, παρουσιάσουμε ε, άλλη μία ε, υποψηφιότητα που έχει μεγάλη εμπειρία στο συνδικαλιστικό κίνημα και νομίζουμε ότι από αυτή την άποψη θα συμβάλλει θετικά στις εργασίες της ε, Επιτροπής. Η Άγνες Λιουγκέριος είναι εδώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, συμφωνεί με την υποψηφιότητά της, έχει υποβάλει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, οπότε αν συμφωνείτε παρακαλώ για την θέση του τέταρτου αντιπροέδρου. Με συγχωρείτε, υπάρχουν άλλες προτάσεις. Όχι. Ωραία, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία Ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η σύσταση σε σώμα της Επιτροπής. Να πω δύο λόγια τότε για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Όπως είπα και εγώ ε, ε, δεν έχω εμπειρία στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θέση. Ήμουν βέβαιος ε, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να εξοικειωθώ κι εγώ με τις ε, εργασίες. Να σας πω δύο λόγια πρωτού ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή έχει να αντιμετωπίσει σε ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες προκλήσεις. Ε, η αναργία είναι στην Ευρώπη πολύ ψηλή βρίσκεται σε πτωτική τάση, ωστόσο το 10,4 εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ψηλό ε, ποσοστό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα είναι και η νεανική ε, ανεργία και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Σε πολλές περιφέρειες και σε κάποιες, ε, σε κάποια κράτη μέλη η νεανική ανεργία προσεγγίζει το 50% ή και υπερβάνει το 50% και αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά η επισφαλής εργασία, εργασία δηλαδή από την οποία δεν μπορεί κανείς να βιοποριστεί, να ζήσει και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας έχουμε στην Ευρώπη περίπου 25 εκατομμύρια εργαζόμενους που ζουν κάτω ή στο όριο της φτώχειας. Νομίζω ότι αυτή η πρόκληση είναι ε, πολύ σημαντική για την ε, κοινωνική, ε, για τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ευρώπης. Στην προηγούμενη θητεία ασχοληθήκαμε με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην Ευρώπη έχουμε ε, πολλές ε, διαφορές όσον αφορά τις σχέσεις εργασίας μόνιμους, μόνιμους και σταθερούς απασχολούμενους, εποχικούς απασχολούμενους, απασχολούμενους με ορισμένο χρόνο. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να ασχοληθούμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι το σύνθημα ίση αμοιβή για ίση εργασία, για ίσο χρόνο και στον ίδιο τόπο ε, θα είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Ωστόσο, στην έναρξη της θητείας θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε και με ζητήματα που ε, έμειναν εκρεμή από την προηγούμενη θητεία θα πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε ή να συνεχίσουμε ε, εργασίες ε, μελών της ε, προηγούμενης θητείας που δεν ολοκληρώθηκαν. Μιλώ συγκεκριμένα για εκθέσεις όσον αφορά τις προτάσεις νομοθετικές για τους ναυτικούς, για την ανάπτυξη και την απασχόληση και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κύρωση της ε, σύμβασης του IMO, της, Διεθνής, της Διεθνούς Ναυτιλιακής ε, Οργάνωσης. Έχουμε επίσης ε, εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για τον προϋπολογισμό, για ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εγγύων στην, στο χώρο εργασίας και με ζητήματα ε, του προσωπικού εδάφους στα αεροδρόμια. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα πρέπει από την 7η θητεία τελικά να ε, διευθετηθούν στην 8η θητεία και οι ομάδες πιστεύω ότι θα ορίσουν σε έφθετο χρόνο και θα δώσουν στους εισηγητές τους τις ε, κατάλληλες οδηγίες ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες αυτές χωρίς προβλήματα. Οι συντονιστές της ε, Επιτροπής Απασχόλησης θα οριστούν ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία. Οι συντονιστές θα ορίσουν μια σειρά από εισηγητέ για τις εργασίες, ώστε στην διάρκεια της νέας μας θητείας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τα καινούρια θέματα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το Eures, την πλατφόρμα για την καλύτερη ε, συνεργασία και την ε, αποτροπή της μαύρης εργασίας στην Ευρώπη και την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία της υγείας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ξεκινούμε με τις εργασίες της Επιτροπής μας επί Ιταλικής Προεδρίας. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε με την Ιταλική Προεδρία, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της ανεργίας των νέων και η Ιταλία όπως έμαθα, είναι χώρα που πλήττεται από υψηλή ανεργία των νέων και στο πλαίσιο της ε, Ιταλικής Προεδρίας θα ασχοληθούμε με την κοινωνική διάσταση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και στην επόμενη κιόλας συνεδρία της Επιτροπής θα έχουμε την δυνατότητα να ασχοληθούμε με την ουσία ε, του ζητήματος. Θα μας επισκεφτεί ο Ιταλός Υπουργός Εργασίας, ο κ. Στολέτη, ώστε να μπορέσουμε να σχηματίσουμε εικόνα ως Επιτροπή ε, ποιε είναι οι επιδιώξει τη Ιταλική Προεδρία. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή για τι εργασίε τη Επιτροπή μα, ώστε να αποκτήσουμε κατευθείαν μια συγκεκριμένη τριβή όσον αφορά τι ε, επιδιώξει της Ιταλικής Προεδρίας. Επίσης, θα πρέπει σύντομα να καταρτήσουμε το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής μας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε πριν από το διάλειμμα που θα κάνουμε για το καλοκαίρι. Μάλλον όχι, αλλά σε αυτή την περίπτωση σίγουρα στις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει η δυνατότητα να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα ε, κατατεθεί ως προσχέδιο από τους συντονιστές όταν αυτοί οριστούν και στη συνέχεια θα υπερψηφιστεί από την Επιτροπή σε συνεδρίαση ολομέλειας της Επιτροπής. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Να σας ενημερώσω επίσης ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής για το υπόλοιπο του 2014. Βρίσκεται στα έγγραφά σας ένα έγγραφο από την Γραμματεία της Επιτροπής Απασχόλησης. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει στις 22 Εβδόμου εδώ στην, ε, ε, στις Βρυξέλλες από τις 3 το απόγευμα έως τις 6. Τουλάχιστον αυτό βλέπω να γράφει το δικό μου χαρτί εδώ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις όσον αφορά αυτά που είπα. Όχι, από ό,τι φαίνεται, οπότε να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι και να σας ευχηθώ στις ομάδες, που, στις επιτροπές που ε, συμμετέχετε. Καλές εργασίες. Θα τα ξαναπούμε στις 22 Ιουλίου, 3 το απόγευμα. Τέλος συνεδρίας. Okay.